Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ, θα πρέπει να τελειώσουμε αυτή τη διαδικασία ψηφοφοριών μέχρι τις 9.45, διότι οι περισσότεροι από εσά <clears throat> θα πρέπει να πάτε στις συνεδρίες της ομάδας σας. Έχουμε κυρίως τις ψηφοφορίες για τις τροπολογίες που αφορούν το σχέδιο έκθεσης για τη μεταρρύθμιση του πολιετούς ε, ε, δημοσιονομικού πλαισίου στα μέσα του δρόμου. Θα ήθελα να ξέρω αν συμφωνείτε για την ημερησία διάταξη. Να σας υπενθυμίσω ότι το σημείο 7 θα εξεταστεί μεταξύ του σημείου 3 και του σημείου 6 και το σημείο 6 θα πάρει τη θέση του σημείου 4. Το σημείο 9 δεν θα εξεταστεί, θα το αναβάλουμε και θα αναβάλουμε επίσης και τις ψηφοφορίες για τα σημεία 5 καθώς και 8. Με άλλα λόγια, θα εστιάσουμε στη μεταρρύθμιση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και θα εξετάσουμε και τις μεταφορές πιστώσεων. Οι συντονιστές συνεδρίασαν χθες. ενέκριναν την αλλαγή της ε, ημερομηνίας της συνεδρίασης της Επιτροπής μας που προβλεπόταν να γίνει την 1η Σεπτεμβρίου και αυτό επειδή την 1η Σεπτεμβρίου θα γίνει ο τριγωνικός διάλογος για τον προϋπολογισμό του 2017 και διαθεσμικές ε, συναντήσεις για τις πιστώσεις πληρωμών. Οπότε εμείς θα συνεδριάσουμε στις 31 Αυγούστου. Οι συντονιστές έδωσαν εντολή στην γραμματεία μας να προετοιμάσει ένα τεχνικό υπόμνημα για τις ε, δημοσιονομικές συνέπειες του Brexit που θα οδηγήσει και σε τροποποίηση της χρηματοδότησης της ε, Βρετανικής έκπτωσης. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια αξιολόγηση της συνεισφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου, ο υπολογισμός της έκπτωσης και τα κονδύλια, τα, θα πρέπει να υπολογιστούν και τα κονδύλια τα οποία αποδίδονται στο νούμερο Βασίλειο και στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε τις αντισταθμίσεις οι οποίες θα πρέπει να προκύψουμε για τα κράτη-μέλη δεδομένου του γεγονότος ότι το Βρετανικό, η Βρετανική έκπτωση χρηματοδοτείται με ένα ειδικό σύστημα το οποίο δεν ε, με τον ίδιο τρόπο όλα τα κράτη-μέλη. Αυτά ήθελα να σας πω λοιπόν. Σας υπενθυμίζω ότι ο πρόεδρος Σούλτς μας προσεκάλεσε στη διάσκεψη που θα γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου για τους ίδιους πόρους. Θα είναι σημαντικό λοιπόν για την επιτυχία αυτής της συνδιάσκεψης να είμαστε πολύ ε, ως μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών που θα λάβουμε μέρος σε αυτή τη διάσκεψη και που θα συμμετάσχουμε φυσικά στη συζήτηση και ενδεχομένω μπορείτε να εκμεταλλευτείτε και αυτή τη συνάντηση για να έρθετε σε επαφή με τις αντιπροσωπείες που θα έρθουν από τα Εθνικά Κοινοβούλια και έτσι να ενισχύσετε τους ε, δεσμούς μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ερχόμαστε λοιπόν στις προφορίες για την προετοιμασία της ε, αναθεώρησης του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020. Προφανώς θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον Γιάννο Όλμπερτ και την Ιζαμπέλ Τομά, τους δύο εισηγητές μας που έχουν κάνει ένα εξαιρετικό έργο και νομίζω ότι χάρη στο έργο τους θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για αυτήν την μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού πλαισίου. Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο για την εκπόνηση μιας θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τροποποίηση του πλαισίου 2014-2020 επί τη βάση μιας ε, ε, αξιολόγησης των προτάσεων της Κομισιόν. Περιλαμβάνει λοιπόν και προτάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενδιάμεση αναθεώρηση και της απόψη του Κοινοβουλίου για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο επέκεινα του 2020 με τα γεγονότα τα οποία έχουν λάβει χώρα με το δημοψήφισμα που οδήγησε στο Brexit έχουμε και μια ουσιαστική και αποφασιστική στιγμή για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης και για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας υπενθυμίζω ότι η συζήτηση για την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2015 επί βάση ενό εγγράφου εργασία των δύο συνεισηγητών που καθόρισε το πλαίσιο των προπαρασκευαστικών εργασιών για την μεταρρύθμιση. Υπήρξαν ομάδες παρακολούθησης που οργανώθηκαν στην αρχή του χρόνου για να αντιμετωπιστεί η αποτελεσματικότητα διαφόρων εργαλείων του προπολογισμού 2014-2020 και των αντιστοίχων <clears throat> προγραμμάτων και έγινε και μια δημόσια ακρόαση για τα θέματα αυτά που έγινε στις 17 Μαρτίου. Και εν τέλει να σας πω ότι έχουμε δείξει ένα, έχουμε δείξει μεγάλη σοφροσύνη γιατί κάναμε ό,τι μπορούμε, ότι μπορούσαμε να μην επηρεάσουμε με την ψηφοφορία μας την ε, ψηφοφορία στο Βρετανικό Δημοψήφισμα γιατί θεωρήσαμε ότι αυτές οι ψηφοφορίες έπρεπε να γίνουν μετά τις 23 Ιουνίου. Θέλω να ευχαριστήσω και τους εκπροσώπους της Κομισιόν για τη συμμετοχή τους στην διαδικασία αυτή και πριν δώσω το λόγο στους εισηγητές θέλω να τονίσω ότι ευχή μου είναι οι προτάσεις της Κομισιόν να λάβουν υπόψη και τις προτάσεις που διατυπώνται στην έκθεση των δύο συνεισηγητών μας. Και δίνω το λόγο πρωτού περάσουμε στις ψηφοφορίες στους δύο εισηγητές. Θέλετε να πείτε κάτι? με την άδειά σας. Εγώ θα προτιμούσα να μιλήσω μετά την ψηφοφορία, λέει η κυρία Τόμα. Εγώ θα μιλήσω πριν. Αντίθετα, λέει ο κύριος Όλμπριχτ, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ε, συντονιστές, τους εισηγητές για το έργο που κάνανε. Είναι ένα πρώτο βήμα. Ξεκινούμε λοιπόν την εργασία για τη μεταρρύθμιση των πολιετών δημοσιονομικών προοπτικών. Αναμένουμε βέβαια τη συνέχεια που θα δώσει η Κομισιόν, αλλά μεταξύ μας έχουμε βρει ικανοποιητικές συμβαστικές λύσεις. Ευχαριστώ επειδή αναφερόσαστε στις ε, συμβαστικές λύσεις, πρέπει να πω <clears throat> ότι μαζί με τους δύο συνεισηγητές έχω διατυπώσει μια τροπολογία που θα σας παρουσιάσω αμέσως και η οποία θα πρέπει να ενσωματωθεί σε μια νέα παράγραφο 28β. Λοιπόν, περνάμε τώρα στη διαδικασία ψηφοφοριών. Παρακαλώ βάλτε τις κάρτες σας για να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ. Θέλω να κάνω μια τεχνική παρατήρηση. Δεν έχω την κάρτα μου εδώ. Κάποιος θα έτοιμασει με την κάρτα μου να μου τη δώσει. Θα έρθει λοιπόν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Παρακαλώ καταγράψτε την ψήφο μου με χειρονακτικό σύστημα. Naturellement, Προφανώς λέει ο πρόεδρος.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 καλύπτεται από τις συμβαστικές 14, 20, 21 αλλά και 22. Επειδή όμως δεν έχουμε φτάσει σε αυτές τις συμβαστικές, ε, τι ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ 15, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 16. Και 17 ταυτίζονται. υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται.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 Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 44. Υπέρ κατά αποχές Απολύτωται 42 υπέρ κατά αποχές <clears throat> Απολύτωται 43 υπέρ κατά αποχές Απολύτωται 45 και 46 που είναι ταυτόσιμες και υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 48 το πρώτο τμήμα μονάχα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο όμως έχει αποσυρθεί. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 50. Υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Αυτό που ψηφίζουμε είναι το χωριστό τμήμα της ε, παραγράφου 50 που έρχεται ως προσθήκη στη Συμβαστική 3. Και είναι λοιπόν προσθήκη στη Συμβαστική 3. Ποιος είναι υπέρ της 50 λοιπόν. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεν λειτουργεί το σύστημα. Έχουμε περιπλέοντες από το ΕΛΚ. Όχι, όχι. Υπάρχει ένας από το ΕΛΚΟ ο οποίο είναι ε, επιπλέον. Λοιπόν, κατάξιστες πώς σας θέσεις πέραση ψηφοφορίες. 18-16, εγκρίνε. 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστή 4 υπέρ. <clears throat> Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 68. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστή 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η 123 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 126 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 131 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 133 και 134 από εκείνο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή 135 εδώ έχουμε πολλά τμήματα. Το πρώτο τμήμα καλύπτεται από τη συμβιβαστική 14. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Το τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τέσσερα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Το πέντε υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Το 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 63. Εδώ για τον τίτλο πάλι δεν ψηφίζουμε. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τέταρτο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το πέμπτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 249 και 251 από κοινό Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτές. 255 υπέρ. Α, για μια στιγμή ε, έχει καταπέσει πλέον γιατί έχουν υιοθετηθεί άλλες. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 141 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές δεκτή 145 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 146 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 149 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 148 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 153 έχει αποσύρθει. 154. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Το δεύτερο τμήμα έχει αποσύρθει. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 159 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 160 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 161 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 163. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 162 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 165 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πρώτη προφορική. Στο 28α. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 168. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Και εδώ υπάρχει και προφορική τροπολογία στην 168. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν. Δεκτή. Και εδώ έρχεται η προφορική με τη σύμφωνη γνώμη του κυρίου Όλμπριχτ. Συμφωνεί η κυρία Τωμά. το 28β του κειμένου. Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει στις αρχές του προϋπολογισμού όλες τις σχετικές πληροφορίες για πιθανές επιπτώσεις σε δημοσιονομικό επίπεδο από τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος χωρίς αυτό να προκαταλαμβάνει την κατάληξη των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέτω σε ψηφοφορία ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν, δεκτή. 167 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 169 υπέρ, Για το 167 θα υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Le scrutin. Le Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 19 υπέρ, 17 κατά. 169. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 170 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 170. Ψηφίζεται. Σκοτά εκλού. Πέρας ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. 19 κατά 17 υπέρ. Καλώς. Συμβιβαστική 18. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 181 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 184 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 185 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 186 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 187 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 188 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 19. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 20. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 211 υπέρ. Κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 212 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 225 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 226 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 224 έχει αποσύρθει. 227. 227 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 227 ψηφίζεται. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 17 υπέρ, 18 υπέρ, 17 κατά. 2,29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 228 υπέρ. Κατά. Α, έχει καταπέσει 228. 230 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 231 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 233 233 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 234 υπέρ κατά αποχές δεκτή 235 υπέρ έχει καταπέσει 2.35, συγγνώμη. Η 236 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 237 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 238 υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. 239 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 240 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 241 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 242 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 243 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 2.44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 2.46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 2.47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστή 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 349. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 27. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 2.66 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28 συμβιβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 281 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 285 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 286 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 290 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 291 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.87 έχει αποσύρθει 2.88 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 294 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 295 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 298 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 300 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 301 υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβιβαστική 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 353 λέει ο πρόεδρος Α, ε, με Προχώρησε πολύ γρήγορα. 308. 308. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 311 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 309 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη 312 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 313 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη. 314 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη. 315 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη. 316 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη. συμμεβαστική 31 υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται. 325 υπέρ. Κατά. Απερίφθη. 326 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 327 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 328 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Συμβιβαστική 32 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 333 υπέρ αποχές εγκρίνεται 335 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 338 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 336 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 337 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 339 υπέρ κατά αποχές Απερίφθη. 343 344 υπέρ κατά αποχές απερίφθησαν Συμβαστική 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 353 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 354 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 355 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, τροπολογία 3 του σκέψη α υπέρ κατά δεν σηκώσατε όλα τα χέρια το επαναλαμβάνω τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 6 ε, υπέρ κατά αποχές απερίφθη 7 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 8 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 9 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 10 υπέρ κατά αποχές απερίφθη υπεριθμόν 1 υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έχουμε επίσης στις νομοδοτήσεις των επιμέρους επιτροπών. Κύριε Όλμπριχτ, θέλετε να πείτε κάτι, οι συγγητές μας έχουν λάβει υπόψη. Ναι, και νομίζω συμφωνεί η κυρία Τωμά. Θέλουμε να υπογραμμίσουμε την πολύ σημαντική συμβολή των επιμέρους επιτροπών. Θελήσαμε να συμπεριλάβουμε τις προτάσεις τους όλες στις συμβαστικές προτάσεις μας. Έτσι λοιπόν καλύπτουμε στις συμβαστικές τροπολογίες όλες τις προτάσεις των επιμέρους επιτροπών. Αυτή είναι η προτάση μας. Καλώς λέει ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριε Ρούμπιχ, Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Έχει λάβει χώρα ένα δημοψήφισμα στο Ρωμανό Βασίλειο. Κάποιοι εδώ έχουν καλέσει σε αποχώρηση από την δημοκρατία την ευρωπαϊκή. Λένε ότι η δημοκρατία σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι αποδεκτή. Εκείνοι λοιπόν οι οποίοι θεωρούν ότι μπορούν να υπόσχονται στο λαό τέτοια πράγματα, νομίζω ότι δεν πρέπει να έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν εδώ μέσα γιατί εδώ έχουν ξεγελάσει το λαό. Ο λαός ψήφισε με το δημοψήφισμα. Δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα να παραμένουν στο κοινοβούλιο και να συμμετέχουν σε ψηφοφορίες. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Μάλιστα. Λαμβάνω γνώση της δηλώσεως σας. θα πρέπει κατόπιν τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματο οι βρετανικέ αρχέ να προβούν στην κοινοποίηση του άρθρου 50 τη συνθήκη. και θα πρέπει να περιμένουμε την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων που θα ξεκινήσουν και που μπορεί να κρατήσουν και δύο χρόνια ακόμη. βεβαίω και το δημοψήφισμα θα έχει ε, συνέπειε για τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα προσπαθήσουμε να προβλέψουμε αναλόγω τι αλλαγέ. Τώρα, σύμφωνα με τις επιθυμίες που εξέφρασαν οι εισηγητές που μας εξήγησε ο κύριος Όλμπριχτ ε, σχετικά με τις γνωμοδοτήσεις των επιμέρους επιτροπών που είναι πολύ σημαντικές και λαμβάνονται υπόψη από τον εισηγητή ε, δεν χρειάζεται να διεξαχθεί για τις γνωμοδοτήσεις αυτές χωριστή ψηφοφορία και έτσι περνάμε στη συνολική ψηφοφορία για το κείμενο ολόκληρο όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. «29 ψήφοι υπέρ, 5 ψήφοι κατά, μία αποχή εγκρίνεται συγχαρητήρια στους εισηγητές μας και σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού έργου και μια και είμαστε σε περίοδο ευχών, εκφράζουμε την ευχή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις προσεχείς ημέρες και εβδομάδες να λάβει γνώση και υπόψη το περιεχόμενο αυτής της τόσο σημαντικής εκθέσεως που θα προσδιορίσει και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μερικά λεπτά ακόμα στη διαθεσή μας και θα παρακαλέσω τον κύριο Ντεπρέ να λάβει το λόγο γιατί έγινε μια συζήτηση για τις πιστώσεις των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Εξωτερικής Δράσης. Θέλουμε κάποιες πληρωματικές πληροφορίες, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ πήρα αυτές τις πληροφορίες και θεωρώ ότι είναι ικανοποιητικού χαρακτήρα. Σας προτείνω λοιπόν να υπερψηφίσουμε την αίτηση αυτή. Ψηφίσουμε με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνονται με 29 έναντι 5 και μία αποχή οι μεταφορές πιστώσεων. Κυρία Τωμά, θέλατε να πείτε κάτι μετά από τις ε, ψηφοφορίες βεβαίως κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα. Απλώς νομίζω ότι έχει σημασία. Θέλω προφανώς να ευχαριστήσω όλους τους συναδέρφους και όλες τις πολιτικές ομάδες που συνέβαλαν όχι μονάχα στο αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας αλλά για την προετοιμασία αυτής της έκθεσης. Θέλω να ευχαριστήσω και εξ βεβαίω του κ. Όλμπρεκ και, του, και εμού της ιδίας της υπηρεσίας του Κοινοβουλίου, τους συνεργάτες μας και τους βοηθούς μας. Θέλω να υπογραμμίσω το θέμα των γνωμοδοτήσεων των ε, επιμέρους επιτροπών. Το είπα και κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Στον προϋπολογισμό <clears throat> δεν μπορούμε να εντάξουμε πολιτικές τομεακού χαρακτήρα. Βλέπω τον κύριο Μαραγκάλ, τον κύριο Μαζί ίσως δεν ικανοποιήθηκαν από όλα αυτά, <clears throat> αλλά δεν μπορούμε στον προϋπολογισμό να αλλάξουμε τις ε, πολιτικές του κάθε τομέα. Λάβαμε υπόψη αυτές τις ε, γνωμοδοτήσεις των Επιτροπών, αλλά δεν μπορούμε να περάσουμε από το παράθυρο αυτό το οποίο δεν μπορεί να μπει από την πόρτα. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω και τους ε, συντάκτες γνωμοδοτήσεων των Επιτροπών για την κατανόησή τους και σας λέω και πάλι ότι είμαστε μονάχα στην απαρχή μιας μακράς πορείας και θα πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε όπως ε, ξεκινήσαμε σήμερα και επειδή είναι πολλά τα διακυβευόμενα θέλω όλους σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και τη συμμετοχή σας. Ναι, λέει και ο και εγώ σας προσκαλώ να κατανοήσετε πόσο σημαντική ήταν αυτή η ψηφοφορία. Ήταν πολύ ευχάριστη αυτή η χρονική στιγμή. Τα επόμενα βήματα ίσως δεν θα είναι τόσο ικανοποιητικά. <clears throat> Ας χαρούμε λοιπόν αυτή τη στιγμή. Θα μας δώσει δύναμη για το μέλλον. Κύριε Ντεπρέ, έχετε κάτι ακόμα για, τα, για τις μεταφορές πιστώσεων από το, του ελεκτικού συνεδρίου. Ναι κύριε Πρόεδρε, το ελεκτικό συνέδριο μας προτείνει τέσσερις μεταφορές πιστώσεων το πρώτο είναι 780.000 ευρώ που αιτιολογείται από το γεγονός ότι είναι απαραίτητο να καλύψουμε το κόστος που προέρχεται από τις αλλαγές των μελών και ιδίως από την αποχώρηση του Προέδρου του Ελεκτικού Συνεδρίου τον Οκτώβριο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεύτερον, 126.000 ευρώ <coughs> για ε, ιατρικές ε, εξετάσεις, αντιμετώπιση ατόμων με ε, αναπηρίες ε, και τα λοιπά και επίσης κονδύλια για την υπηρεσία μετάφρασης λόγω του γεγονότος ότι ο αριθμός των ειδικών εκθέσεων έχει αυξηθεί. Πιστεύω και δεν πρόκειται να αντιδράσω βέβαια σε αυτήν την μεταφορά πιστώσεων, να πρέπει να ζητήσουμε και από το ελεκτικό συνέδριο να μας εξηγήσει πώς επιλέγουν τις ειδικέ εκθέσεις οι οποίες έχουν πολλαπλασιαστεί. Είναι δύσκολο να τις παρακολουθήσει όλες. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να έχουμε και μια σοβαρή συζήτηση με το ελεκτικό συνέδριο για τις εκθέσεις αυτές, αλλά δεν έχω καμία αντίρρηση για αυτή τη μεταφορά πιστώσεων. Τέταρτη μεταφορά, 75.000 ευρώ για το ε, πολυσίδες κέντρο της ε, ε, για τα παιδιά, για, για την παιδική ηλικία, γιατί υπήρξε ανθρωποποίηση στον παιδικό σταθμό. Έχουν υπάρξει προσθήκες παιδιών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, το, και την Κομισιόν και τέταρτη μεταφορά 12.000 ευρώ για την επαγγελματική εκπαίδευση για τα νέα προγράμματα τα οποία θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ηγετική και διαχειριστική ικανότητα. Ε, δεν πρόκειται να πούμε και όχι σε τέτοια προγράμματα, τα οποία θα οδηγήσουν σε τέτοιες ικανότητες. Είναι μικρό το ποσό και ελπίζω ότι τα αποτελέσματα θα είναι στο ύψος των προσδοκιών μας. Και υποστηρίζω αυτή την, ε, την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων. Κύριος Μανκά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ υποστηρίζω όλες αυτές τις μεταφορές πιστώσεων οι οποίες παρουσιάστηκαν από τον κύριο Ντεπρέ για το μέλλον όμως θα πρέπει να συμφωνήσουμε με το ελεκτικό συνέδριο για το εξή. Το 2006 κάνανε μία έκθεση και λένε ότι αν ένα θεσμικό όργανο δεν έχει ικανότητα για να κάνει περισσότερες ε, μεταφράσεις intramuros θα πρέπει να αναζητήσει και ικανότητα μετάφρασης από εξωτερικούς συνεργάτες. Αν το κάνουμε αυτό όμως θα μπορέσουμε να κάνουμε και εξοικονόμηση χρημάτων. Αλλά το κάνει το ίδιο το ελεκτικό συνέδριο. Πριν ε, κάνουν μεταφράσεις εξωτερικές θα πρέπει να δουν αν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να καλύψουν αυτό. Δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο. Λοιπόν, θα αποφασίσουμε. Εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις, νομίζω ότι μπορούμε να εγκρίνουμε τις πιστώσεις δεδομένου του χαμηλού ποσού. Και δίνω και πάλι το λόγο στον Γενικό Εισηγητή για το τμήμα 3 του προϋπολογισμού 2017, τον κύριο Φερνάντης. 2016, συγγνώμη, 2017 Κύριε Πρόεδρε, και εγώ προτείνω να ε, υπερψηφίσουμε τη μεταφορά 11, 8,8 εκατομμύρια ευρώ, αφορά διοικητικέ ταπάνες για εξωτερικό προσωπικό για δραστηριότητε που έχουν εξωτερικευθεί. Πρόκειται για αναδιάταξη σε ορισμένε γενικές διευθύνσει, οι οποίες έχουν μεγαλύτερο φόρτο εργασία και ιδίω στη Γενική Διεύθυνση που έχει να κάνει με την αντιμετώπιση τη κρίση των, της και μεταφορές από την Ντέτζε Ρέζιο Κέφα προς τη Γενική Γραμματεία. Η πρότασή μου λοιπόν είναι να υπερψηφίσουμε αυτές τις μεταφορές πιστώσεων. Ωραία λέει ο πρόεδρος. Με ονομαστική κλίση λοιπόν άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. οι μεταφορές πιστώσεων έχουν εγκριθεί. Και ερχόμαστε στην έκθεση Γκάια για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία <clears throat> Εναέρειας Ασφάλειας. Ζητώ από τον κύριο Μουρεσάν να αναλάβει την Προεδρία, γιατί είμαι υποχρεωμένος να φύγω. Και σας ζητώ συγγνώμη που πρέπει να φύγω. Παρακαλώ. Ερχόμαστε στην ψηφοφορία για την έκθεση του κυρίου Γιανσκάια για τον τομέα της ε, ε, υπηρεσίας αεροπορικής ασφάλειας. Η πρότασή μου είναι για τις τροπολογίες 28-37 να ψηφίσουμε unblock. Συμφωνείτε? Ψηφίζουμε λοιπόν τις τροπολογίες 27, 28-37 από κοινού σε ψηφοφορία. Παρακαλώ. Κύριε Τσάνη, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ζητήσω να ψηφίσουμε ξεχωριστά, μεμονωμένα, γιατί θέλω να ψηφίσω με διαφορετικό τρόπο. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε ομαδών. Καλώς θέτουμε λοιπόν την 28 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, αποχές, απορρίπτεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 ποιοι είναι υπέρ κατά Νομίζω ότι θα υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 38 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 21 υπέρ 11 κατά. 39 υπέρ κατά. Αποχές. Δεκτή. 40 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 41 μέχρι 67. Θα κάνω την ίδια πρόταση να ψηφίσουμε ομαδών. Από την 41 μέχρι την 60. Μέχρι την 60. Μπορούμε παρακαλώ όλες μαζί. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τίθενται σε ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Περνάμε τώρα. Την 61. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία υπάρχουν 3 Πέραση της ψηφοφορίας. Δεκτή. 18 υπέρ, 17 κατά. Τροπολογία 4. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η ίδια πλειοψηφία. 5. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 68 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 69 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Θα υπάρξει έλεγχος ηλεκτρονικός λοιπόν για την 6. Ψηφίζεται. Πέρας ψηφοφορίας. 19 υπέρ, 16 κατά. Δεκτή. Η 70 έχει καταπέσει. Η 7 τώρα, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της 7. Ψηφίζεται. Τέλος. 19 υπέρ 16 κατά. Δεκτή. Η 71 έχει αποσυρθεί. Η 72 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για την 8. Ψηφίζεται. Τέλος. Δεκαεννέα υπέρ, 16 κατά. Εννέα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Αυτό σημαίνει ότι έχει καταπέσει 73. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά κατά, αποχές, δεκτή. 17 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1 υπέρ, κατά, αποχές, Ηλεκτρονικός έλεγχος για την πρώτη τροπολογία. Ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφη. Τροπολογία 22. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 22. Ψηφίζεται. Τέλος, απερίφη. 23 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφη. 24 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφη. 2 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφη. Αυτό σημαίνει ότι ψηφίζουμε τώρα την 25. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή 26 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 27 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 74 υπέρ κατά αποχές δεκτή τώρα το σύνολο με ηλεκτρονική ψήφο ψηφίζεται πέρας ψηφοφορίας η έκθεση απερίφθη. Έχει απορριφθεί η έκθεση. Περνάμε τώρα στην επόμενη έκθεση. 16 υπέρ, 16 κατά, δεν αλλάζει το αποτέλεσμα, έχει απορριφθεί η έκθεση. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα, στην ημερήσια διάταξη. Έκθεση Μούντι. Ψηφίζουμε τώρα τη συμβοβαστική α. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Συμβιβαστική α, ηλεκτρονικός έλεγχος ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή, 18 υπέρ, 17 κατά. Οπότε δεν ψηφίζουμε εφόσον έγινε δεκτή η συμβιβαστική α. Η 2 καλύπτεται, η 1 καλύπτεται. Πηγαίνουμε στην 7 παρακαλώ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Συμβιβαστική β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 12. Ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 13. Υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή 19 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 18 υπέρ Η 19 έχει απορριφθεί, εν πάση και ψηφίζουμε τη 18. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Κοιτάξτε, ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 18, παρακαλώ, ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 18 υπέρ, 16 κατά. Αυτό σημαίνει ότι ψηφίζουμε τώρα ή μάλλον η 17 έχει καταπέσει γιατί έγινε δεκτή η 18. Ψηφίζουμε λοιπόν την 20. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 21 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 21. Τέλος γίνεται δεκτή 18 υπέρ 14 κατά 22 υπέρ κατά αποχές απερίφη η 23 έχει πλέον καταπέσει ψηφίζουμε την 24 με προφορική τροπολογία του εισηγητή ποιοι είναι υπέρ ποιοι είναι κατά αποχές 25 υπέρ κατά αποχές απερίφη 26 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική C αγγλικό, υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν για τη συμβιβαστική C. Τέλος ψηφοφορίας, 18 υπέρ, 17 κατά. Περνάμε τώρα στην 32, ποιοι είναι υπέρ Ζητώ συγγνώμη λέει ο Πρόεδρος. Την 28 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Τώρα θα ψηφίσουμε την 32 υπέρ, κατά, ηλεκτρονικό ηλεκτρονικός έλεγχος για την 32. Ψηφίζεται. «20 υπέρ 14 κατά» το σύνολο του, της νομοδότησης όπως τροπολογήθηκε. Ψηφίζεται. Τέλος. 30 υπέρ, 2 κατά και 3 αποχές. Ευχαριστώ πολύ. So, um, um, so are we doing transfers or? No, there's none. Um, as, as the time for, uh, there are, Ms. Holmeyer, are there any... Κυρία Χολμάιερ, υπάρχουν μεταφορές αυτή τη φορά. Όχι. Δεν υπάρχουν λοιπόν μεταφορές, δεν υπάρχουν άλλα θέματα. Τέλος της συνεδρίασης, η επόμενη συνεδρίασή μας την 30 Ιουνίου. Ευχαριστώ.